Ευρώπη προς το συμφέρον των Μολδαβών πολιτών και της Ευρώπης επίσης. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Έχουν υποβληθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος για την ολοκλήρωση της συζήτησης. Μία από το ΕΛΚ, μία από τους φιλελεύθερους, άλλη πρόταση από την ΚΟΕ, ψήφισμα από τους Περασίνους τους σοσιαλιστές και τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Έξι προτάσεις ψηφίσματος συνολικά και θα τις ψηφίσουμε σήμερα το μεσημέρι. Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα και τη σχετική αποζημίωση. Πρόκειται για μια προφορική ερώτηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Θα την υποβάλει για πέντε λεπτά ο συντάκτης της προφορικής ερώτησης, ο κύριος Σίμψον. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Επιτροπή Μεταφορών για ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε παραβλέψει εδώ και καιρό, δηλαδή τα κοντέινερ που πέφτουν από πλοία στη θάλασσα είναι εκπληκτικό για εμένα, σήμερα ημέρα, χιλιάδες τέτοια είναι να χάνονται κάθε χρόνο και η μεγάλη τους πλειοψηφία πέφτει από τα πλοία στους ωκεανούς. Υπολογίζεται, κύριε Πρόεδρε, πως 10.000 τέτοια εμπορευματοκιβώτια χάνονται στη θάλασσα κάθε χρόνο. Και φαίνεται πως και οι ασφαλιστικέ εταιρείε ε, και οι εφοπλιστικέ εταιρείε αποδέχονται αυτό το νούμερο και δεν κάνουν τίποτα. Στα ευρωπαϊκά ύδατα χάνονται 2.000 κοντέινερ στη θάλασσα, ένα νούμερο που αυξάνεται χρόνο το χρόνο. Αποτελούν απειλή για την αυσιπλοεία, θα μπορούσαν να μολύνουν τις θάλασσες με τοξικά και μη τοξικά υλικά και επιβαρύνουν και τις τοπικές αρχές με το κόστος καθαρισμού. Η Επιτροπή Μεταφορών τώρα ζητά δράση για να μειωθεί αυτός ο αριθμός και στέλνει ένα μήνυμα στην αυτιλιακή κοινότητα πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση για πολύ περαιτέρω. Το Ινστιτούτο Μαρίν, το Θαλάσσιο Ινστιτούτο της ε, Ολλανδίας ε, ανακάλυψε πως ε, το πρόβλημα αυτό οφείλεται σε λάθος πρόσδεση και αποθήκευση. Επιπλέον, το πλήρωμα στα μεγαλύτερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων έχουν πρόβλημα να αξιολογήσουν το ότι γίνεται με τα τελείως ακραία κυβότια, ειδικά όταν υπάρχουν μεγάλες κάθετες επιταχύνσεις που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές του πλοίου. Επιπλέον, το ότι δεν υπάρχει μια αυστηρή σύμβαση για, αστική, για αποζημίωση αστική ευθύνη για μη τοξικέ ε, ουσίες ε, σημαίνει πως επιβαρύνονται οι τοπικές αρχές με τον καθαρισμό. Αυτό το οποίο ζητάει τώρα το Κοινοβούλιο είναι οι ναυτιλιακές εταιρείε να αποδεχθούν τις ευθύνες τους και θα θέλαμε η Κομισιόν να δράσει περισσότερο προληπτικά για να αντιμετωπίσει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Ζητάω σήμερα από την Κομισιόν να μελετήσει τα αποτελέσματα του σχετικού έργου για να δει τι γίνεται με τις σχετικές διαδικασίες πρόσδεσης στα πλοία. Τέλος, θα θέλαμε να ζυγίζονται όλα τα κοντέινερ σωστά στα λιμάνια και να αποθηκεύονται σωστά να στηβάζονται σωστά στο πλοίο πριν αυτό αναχωρήσει, καθώς και να αποκτήσουν όλα αποδέκτες για να μεταδίδουν τη θέση τους. Και τρίτον, ζητάμε από την Κομισιόν να εξετάσει το καθεστώς αποζημίωσης, έτσι ώστε τοπικές και περιφερειακές αρχές να μην καταλήγουν να πληρώνουν τη ζημιά. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στις υποχρεώσεις ε, τομέα της ναυτιλίας. Εκτιμώ πως όταν, είναι, όταν έχουμε σοβαρές θύελες θα χαθούν κάποια κοντέινερ. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι να χάνονται λόγω τσαπατσουλιάς ή να στηβάζονται με λανθασμένο τρόπο ή λόγω μιας χαλαρής αντιμετώπισης από τον κλάδο γενικότερα. Το να πέφτουν κοντέινερ από τα πλοία είναι κάτι επικίνδυνο το να χάνονται 20.000 από αυτά το χρόνο είναι απαράδεκτο. Κινδυνεύουν ζωές, γι' αυτό ζητάμε και απαιτούμε δράση. Η ναυτιλία φαίνεται πως δεν θέλει να δράσει. Ίσως θα έπρεπε να δράσουμε εμείς κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απαντήσει ο Επίτροπος Γκέγκαν Κουίν. Ε, Κύριε Επίτροπο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σίμψον γιατί είναι πολύ σημαντική η προφορική του ερώτηση και ενδιαφέρει πολλούς ευρωβουλευτές. Νομίζω ότι το θέμα αυτό αφορά κυρίως τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ε, που ασχολείται με τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα, γιατί οι ρυθμίσει ε, αποφασίζονται διεθνώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να προωθήσει δράσει προκειμένου να υλοποιηθούν οι διεθνεί συμφωνίε στα πλαίσια του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού. Σε ό,τι αφορά το υπέρβαρο και το κοντέινερ που δεν έχουν ε, αποθηκευτεί σωστά, δεν υπάρχουν κοινοτικέ διατάξει που να διέπουν τον τρόπο αποθήκευση των εμπορευματοκιβωτίων. Είναι θέμα εθνικό ή διέπεται από διεθνείς συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Βέβαια, η κατάσταση θα μπορούσε να ανάξει αν δεν τελεσφορήσουν οι διεθνείς συζητήσεις και ενισχυθούν τα προβλήματα αυτά εξαιτία τη αστάθεια πλοίων ή υπερβολική απώλεια πορευματοκιβωτίων. Φυσικά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε τον αντίκτυπο ενό τέτοιου μέτρου σε, εφο, σε εφοπλιστικέ εταιρείε. Θα πρέπει επίση ε, για το τρίτο θέμα, για το θέμα της ανείχνευσης και εντοπισμού των εμπορευματοκιβωτίων. Αυτό θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Βέβαια, θα ήταν πολύ δαπανηρή η διαδικασία εξοπλισμού των εμπορευματοκιβωτίων με συσκευέ που θα, θα επιτρέπουν τον εντοπισμό τους και θα ήταν ίσως ε, πολύ επαχθές να γίνει δεσμευτικό ένα τέτοιο σύστημα. Ε, έχουμε και την οδηγία 59 του 2002 που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο, πλοιο, ο ε, κυβέρνητης του πλοίου θα πρέπει να ενημερώνει για τον αριθμό και το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων που χάνονται στη θάλασσα. Βέβαια, μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να εξεταστεί στα πλαίσια των ε, μελλοντικών εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ανιχνευσιμότητα για λόγους ασφάλειας των ε, κοντέινερ. Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση, από τα χαμένα εμπορευματοκιβώτια. Εδώ η οδηγία 2009-20 θα μπορούσε ίσως ε, να ισχύσει και επίσης η οδηγία 2005-35 για την ε, ρήπανση της θάλασσας και τις κυρώσεις. Ε, εκεί καλύπτονται οι περιπτώσεις που ε, πραγματοκιβώτια με πετρέλαιο έχουν χαθεί στη θάλασσα. Και η οδηγία 2004-35 προβλέπει σημαντική ευθύνη για παρόχους που ρηπαίνουν το περιβάλλον εξαιτίας θαλάσσιας μεταφοράς επικίνδυνων ή ρηπογόνων αγαθών. Τέτοιου είδους πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να διορθώσουν τη ζημία που έχει προκληθεί στο οικοσύστημα ή σε διάφορα είδη. Και υπάρχει και καθεστώς αποζημίωσης θα πρέπει όμως αυτό να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας που θα πρέπει να δικαιολογεί τις κοινοτικές δράσεις. Αυτή τη στιγμή το έργο του Διεθνούς Νεοφυλακού Οργανισμού για τη βελτίωση των προδιαγραφών και των προτύπων είναι κατά τη γνώμη μας η σημαντικότερη προτεραιότητα. Ευχαριστώ εκ μέρου των ομιλητών των ομάδων. Θα ακούσουμε πρώτα για δύο λεπτά τον κύριο Ρικέ εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όπως υπενθύμησε ο κύριος ε, Λί ε, Σίμψον, ε, χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια χάνονται στη θάλασσα και είναι πρόβλημα καταρχάς για λόγους μόλυνσης, το οποίο αναφέρθηκε παρκώς, αλλά και γιατί πολλά από αυτά δεν βουλιάζουν και επιπλέον δεν είναι εύκολο να τα εντοπίσουμε και αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και των, εμπορευμα... των ε, εμπορικών πλοίων, αλλά και για τα σκάφη αναψυχής. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν γίνει σοβαρότατα ατυχήματα ε, με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Είναι ένα τεράστιο λοιπόν πρόβλημα και θα ήθελα η Κομισιόν να μας απαντήσει, να μας πει ας πούμε ότι δεν έχει πληροφορίες για να δράσει ή θεωρεί ότι με βάση το σημερινό πλαίσιο και διατάξεις ε, προβλέπονται κάποια πράγματα, κάποια μέτρα ε, και δεν είμαστε εντελώς ε, στερημένοι εργαλείων. Εγώ θέλω να προταθούν αποτελεσματικά μέτρα και προληπτικά, δηλαδή για τους τρόπους ε, φόρτωσης και πρόσδεσης των εμπορευματοκιβωτίων και δεύτερον για την δυνατότητα, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με οικονομικό τρόπο, ε, ανείχνευσης των εμπορευματοκιβωτίων που επιτρέπει από τη μία να τα εντοπίσουμε όταν χάνονται ή να τα αποφύγουμε όταν ή επίσης να τα ανακτήσουμε σε περίπτωση που περιέχουν τοξικά προϊόντα. Θα πρέπει αυτά τα, αυτοί οι ανιχνευτές να εντοπίζουν τα τοξικά ή επικίνδυνα προϊόντα με με ένα μήνυμα ε, ούτως ώστε να προλάβουμε ή να περιορίσουμε τον ε, περιβαλλοντικό κίνδυνο. Επίσης, θα πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε χάρη στην ανείχνευση τον ιδιοκτήτη, γιατί υπάρχει ένα θέμα ευθύνη, το οποίο αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της προφορικής ερώτησης. Η απουσία αναγνωρισμένης ιδιοκτησίας, η ικανότητα εντοπισμού των εμπορευματοκιβωτίων έχει ως αποτέλεσμα ότι και για την ανακτησή τους και για την αποζημίωση δεν προβλέπεται τίποτα. Ζητάμε λοιπόν στεναρά από την Κομισιόν να μην περιοριστεί στο να διαπιστώσει ότι δεν έχουμε τα μέσα να κάνουμε τίποτα ή ότι τα ε, σημερινά μέσα αρκούν. Δεν αρκούν. Υπάρχει θέμα περιβαλλοντικής ασφάλειας, αλλά υπάρχει και θέμα ανθρώπινων ζώων που διακυβεύονται εξαιτία των ε, κοντέινερ αυτών. Για 1,5 λεπτά εκ μέρου των Σοσιαλιστών το λόγο έχει ο κύριο Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, ο Μπράιαν Σίμψον. Η απώλεια κοντέινερ και του περιεχομένου τους, βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτό είναι το θέμα, είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει εκτιμηθεί αρκετά αλλά όπως είπαμε αφορά μόνο στα ευρωπαϊκά ύδατα 2.000 κοντέινερ το χρόνο με συνέπειες για το περιβάλλον και πιθανώς για τους ανθρώπους, για τα άλλα σκάφη, για τις παράκτιες περιοχές και βεβαίω με εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την αποκομιδή τους. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την στίβαση και την πρόσδεση των κοντέινερ. Βεβαίως θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρωτοβουλία. Δεν πρέπει να περιμένουμε παθητικά να λάβει μέτρα ο Διεθνής Οργανισμός Αυτιλίας. Πρέπει να κινητοποιηθούν και να ενημερωθούν τα ευρωπαϊκά λιμάνια και νομίζω πως σε έναν διάλογο με τον ευρωπαϊκό λιμενικό τομέα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθεί σε μια λύση. Τώρα, όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των κοντέινερ, όπως είπε η συνάδελφος, Νομίζω πως είναι σημαντικό όχι μόνο σε σχέση με αυτό το θέμα, αλλά στο όλο πλαίσιο της αλυσίδας επιμελητίας. Και αναμένω βεβαίω του επόμενου μήνε και χρόνια μια πρωτοβουλία από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, το λόγο έχει η κυρία Μάισνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Βλέπουμε τίτλους πως ε, έφτασε ένα φορτίο παπουτσιών ε, σε ένα νησί και χάρηκαν πάρα πολύ οι κάτοικοι του νησιού ή ένα άλλο το οποίο ήταν γεμάτο πλαστικά παπάκια. Αυτέ είναι ευχάριστε περιπτώσεις, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουμε σοβαρές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τα χαμένα αυτά κοντέινερ. Οπότε είναι σαφές το τι πρέπει να κάνουμε. Η Ολλανδική κυβέρνηση ερεύνησε το θέμα, να δει γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αναφέρθηκαν κάποιοι λόγοι, αφενός παρατηρήσαμε πως ε, Υπάρχουν ήδη ευρωπαϊκές ε, διατάξεις για το πώς θα πρέπει να φορτώνονται τα κοντέινερ, οπότε δεν χρειαζόμαστε νέους ε, κανόνες. Αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο ένα 46% των φορτίων ε, στηβάζεται σωστά. Επίσης ε, πάρα πολλά πλοία, ειδικά όταν είναι μικρές οι αποστάσεις, απασφαλίζουν το φορτίο πλην φτάσουν στο λιμάνι για να είναι έτοιμα να ξεφορτώσουν. Και βεβαίως αυτό οδηγεί στο ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλη επιβάλληση του περιβάλλοντος. Ξέρετε πως ένα 70% των ε, απορρίψεων ε, από πλοία βυθίζεται και ένα 15% επιπλέει και άλλο ένα 15% φτάνει στι ακτές. Το 15% που επιπλέει βεβαίω είναι ακριβώς το επικίνδυνο και το ρηπογόνο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα κοντέινερ σε αυτή την περίπτωση, να μιλήσουμε οπωσδήποτε με τους εφοπλιστές και με τα λιμάνια για να εφαρμόσουν τις σχετικές ε, διατάξεις και βεβαίως να υπάρχουν και τακτική έλεγχη. Είναι πάρα πολλά τα 2.000 ε, κοντέινερ. Θα πρέπει να γίνει ε, κάτι. Οπωσδήποτε δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Η κυρία Πάσκα. Ε, ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η λύση της ε, αποζημίωσης ε, από χαμένα εμπορευματοκιβώτια υπάγεται στο τρίγωνο μεταξύ ιδιοκτήτη των εμπορευματοκιβωτίων ε, μεταφορικής εταιρεία και ασφαλιστικής εταιρεία. Βέβαια, τις περισσότερες φορές επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης αλλά και το προσωπικό του πλοίου είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων, την ασφαλή προσδεσή τους και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας για τη μεταφορά αγαθών μέσω θαλάσσης. Είναι πολλές οι αυτού του θέματος και θα πρέπει να βελτιώσουμε τους ελέγχους για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται δια θαλάσσης θα πρέπει να εξετάσουμε και εναλλακτικέ λύσεις για τη μεταφορά αγαθών και την σωστή ασφάλειά τους. Θα πρέπει μόνο, πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε αν όντω ε, οι διατάξεις εφαρμόζονται στην πράξη και να δούμε αν χρειάζονται άλλες ή αρκούν αυτές που δεν εφαρμόζονται όμως σωστά. Σας ευχαριστούμε κύριε Πάσκα. Επόμενος ο ε, από ο κύριος Higgins έχω ολοκληρώσει τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Brian Simpson έθεσε ένα κέριο ζήτημα με την προφορική του ερώτηση και σας διαβεβαιώ ότι είμαι δυσαρεστημένος με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να αναλάβει καμία πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την καλύτερη βελτίωση, την βελτίωση αυτής της κατάστασης και τη διόρθωση. Αν κοιτάξουμε τα στατιστικά στοιχεία, η κατάσταση είναι ακόμη πιο σοβαρή. Περίπου 50% των ε, εμπορευμάτων που μεταφέρονται ε, αχάνονται ε, στη θάλασσα. Επίσης, έχουμε από 32,6% στα 76% το, οι τόνοι που χάνονται τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε την κατάσταση. Υπάρχει το θέμα της αυξανόμενης ταχύτητα, γιατί τα φορτηγά αυτά που, που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια ταξιδεύουν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Ε, εφαρμόζουν μέχρι και 27 ναυτικού κόμβου που είναι πολύ μεγάλη... Ε, ταχύτητα σε σχέση με τον κίνδυνο που υπάρχει, ακόμη και για συγκρούσεις. Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το, την ηλικία των πλοίων. Αν κοιτάξουμε την ηλικία των πλοίων που μεταφέρουν από ρευματοκιβώτη, τα περισσότερα πλοία είναι 90-94 ετών. με 24 ετών. Θα είναι μεγάλες ηλικίες δηλαδή αυτά τα πλοία. Ε, θα πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση και επίσης ε, σημαντικές ε, συμβάσεις για την ασφάλεια, ώστε όταν ε, τα πλοία αυτά μεταφέρονται στα χωρικά κυκλοφορούν στα, χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τηρούνται οι προδιαγραφές της. Σίγουρα χρειάζεται δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται και όπως είπε ο κύριος Σίμψον, τις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ανθρώπινο λάθος αυτό που προκαλεί την απώλεια, το κακή πρόσδεση, η κακή αποθήκευση Γι' αυτό χρειάζονται οπωσδήποτε μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Χίγκινς. Για 1,5 λεπτό η κυρία Γιαλασέντερ. Ευχαριστώ. Τον επόμενο Νοέμβριο θα συμπληρώσουμε 8 χρόνια από, την, από το ναυάγιο του Πρεστίζ στις ακτές ε, της Γαλλικίας που δημιούργησε μια τεράστια ε, πετρελαιοκυλίδα εξαιτίας των αποφάσεων εν μέρη και του, του Υπουργού Κάσκος που δημιούργησε τεράστια οικολογική καταστροφή στις ακτές της Γαλλικίας. Μάλιστα, ένα από τα προβλήματα που οδήγησαν στο ναυάγιο ήταν τα εμπορευματοκιβώτια που επέπλεαν στη θάλασσα και που πραγματικά είναι τορπίλες για ε, για εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία, ακόμη και πλοία αναψυχής. Υπήρξαν τεράστιες αμέλειες σε πολλούς τομείς, στην κατάρτιση και την εκπαίδευση του προσωπικού, αυτούς που στήβαζαν τα, πλοία, τα στα λιμάνια, αλλά και την ελληπή κατάρτιση των πλοηγών. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι τακτικές και για την ειχνηλασιμότητα των βοτιών αλλά να ελεγχθεί και το θέμα του υπέρβαρου. Θα πρέπει να γίνει και μια εκτίμηση κόστους σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτών των τεράτων της θάλασσας. Ίσως θα μπορούσαμε να ελέγξουμε και το πρόβλημα της ε, απώλειας των εμπορευματοκιβωτίων και χρειάζονται και προληπτικά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερη κατάρτιση των ε, ε, λιμενεργατών που στηβάζουν τα πλοία. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και στα λιμάνια για τον έλεγχο, αλλά και να εφοδιαστούν με συσκευέ τα εμπορευματοκιβώτια για να ανοιχνεύονται σε περίπτωση απώλεια. Γιατί η χνηλασιμότητά του ήταν ίσω μία από τι υπηρεσίε του προγράμματο Γαλιλαίο. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα Σέντερ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους πως ε, δεν είναι σωστό να διαβάζετε τους ε, λόγους με τόσο υψηλή ταχύτητα και αν είναι να διαβάζετε ομιλίες από μέσα ε, να σας υπενθυμίσω πως υπάρχει δυνατότητα να τις δώσετε από πριν στους διερμηνείς για να κάνουν και αυτοί κάπως καλύτερη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Λάχιτ φρίτη κατόπιν για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να το λάβω απόψη αυτό που είπατε. Χαίρομαι. για το ότι τον 15ο αιώνα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν υπήρχε ο Κολόμβος και οι φίλοι του θα πέφταν πάνω σε κάνα κοντέινερ και θα βυθίζονταν και δεν θα φτάνουν ποτέ στην Αμερική. Ξέρουμε ποιος στέγει για αυτό το πρόβλημα. Ξέρουμε πως πρέπει να γίνει κάτι. Και τι μας λέει η Κομισιόν, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Δεν είναι σωστό αυτό. Όταν ξέρουμε πως θέλει η λάθος αποθήκευση, όταν λέει πως ε, έχει... Όταν γνωρίζουμε πως είναι υπερφορτωμένο ένα πλοίο και ξέρουμε πως κανένα κράτος δεν μπορεί μόνο του να κάνει κανονισμούς για να το αλλάξει, τότε τι άλλο πρέπει να περιμένουμε για να κινητοποιηθεί η Κομισιόν που υποτίθεται ότι φροντίζει το περιβάλλον στις θάλασσες. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και οι ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν. Εάν ε, ένα σκάφος ε, πολύ ιστερικό ή οτιδήποτε ε, πέσει πάνω σε ένα τέτοιο ε, κοντέινερ. Δεν είναι πολύ αστείο να πέσει κανείς με το σωσίβιο στο Βόρειο Ατλαντικό. Γι' αυτό είναι λάθος το να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να οδηγηθούμε σε αυστηρές σε αυστηρούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Είναι σοβαρή υπόθεση, επικίνδυνη και πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια επιτέλους. Ευχαριστώ κύριε Λάιχτφριντ. Ακριβώς στην ώρα σας περνάμε στη διαδικασία και έτσι ΔΙΑΗ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν το λόγο έχει η κυρία Πυρίλιο. Συγγνώμη, ο κύριος Πυρίλιο. Πρόεδρε. Α, δεν φωνή Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η ερώτηση για τα ε, εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα για την οικονομία των παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί ούτω ώστε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν ε, με αποζημιώσεις ε, οι ζημιές που προκαλούνται από αυτά τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή ναυσιπλοεία με νομοθετήματα πολύ πιο αυστηρά, ε, ελέγχοντας το, τις επιχειρήσεις φόρτωσης-εκφόρτωσης των αγαθών, ειδικά όταν αυτά είναι τοξικά και επικίνδυνα και ρηπογόνα. Ε, τέτοιου τύπου πράγματα τα έχω ζητήσει σε ανάλογες ε, συζητήσεις, σε ανάλογες υποθέσεις. Ζητάω κυρίως ένα καθεστώς ε, αποζημίωσης. Ευχαριστώ. Η διαδικασία και έτσι θα ολοκληρωθεί με τον κύριο Σίμψον. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο και να πω πω απογοητεύτηκα από την απάντηση της Κομισιόν στο προφορικό μας ερώτημα. Αντιλαμβάνομαι πως το ιδιώδες θα ήταν μια παγκόσμια συμφωνία και πως πρέπει να εμπλακεί ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, αλλά ο IMO πραγματικά πρέπει να είναι ένας από τους πιο αργοκίνητους ε, διεθνείς οργανισμούς. Κινείται με ρυθμό χελώνας και εμείς θέλουμε να δράσουμε τώρα. Κυρία Πρόεδρε, εάν εγώ ρίξω 2.000 μεταλλικά κουτιά στη θάλασσα εσκεμένα θα οδηγηθώ στα δικαστήρια. Το επιτρέπουμε όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνω έκκληση. Δεν μπορείτε να παίζετε τον πόντιο πιλάτο και να λέτε νύπτω τα σχήρας μου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αυξάνεται, σοβαρό πρόβλημα και είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσετε. Δεν μπορείτε εδώ πέρα να κρυφτείτε πίσω από τις λέξεις και να λέτε πρέπει να αξιολογήσουμε και δεν ξέρω και εγώ τι. Ακούσατε τι είπαν οι συνάδελφοι. Προσπαθήστε λοιπόν να κάνετε κάτι. Ευχαριστούμε κύριε Σίμψον. Θα ολοκληρώσει η συζήτηση η κυρία Κέικεν Κουίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Και καταλαβαίνω την σημασία της ε, συζήτησης που κάνουμε σήμερα. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προσπαθήσει και αυτή ούτω ώστε να δημιουργήσει μια πολιτική για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι η συζήτηση δείχνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε πως είναι θέμα προστασίας ε, του περιβάλλοντος. Ακούσαμε Ε, διάφορα πράγματα από αυτά που είπε η κυρία Μάισνερ μέχρι τον Κολόμβο που ανέφερε κάποιος ε, βουλευτής. Ε, Κάποιο είπε ότι στη Δυτική Ιρλανδία έφτασε ο Κολόμβος το δικό μου το χωριό. Ε, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη που έκανε το διάσημο ταξίδι του, αλλά θέλω να σας τονίσω ακόμα μια φορά σε όλους και κυρίω σε εσά κύριε Σίμψον, που σας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το θέμα και που έχετε δουλέψει τόσο πολύ γι' αυτό ότι είμαστε σοβαρότατοι για το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε τον μεγάλο αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων που χάνονται και που αυξάνεται μάλιστα αυτός ο αριθμός και μάλιστα θέλω να σας πω ότι ο Αντιπρόεδρος Κάλλας εξετάζει αυτό το πρόβλημα και πιστεύουμε ότι δεν συνδέεται μόνο με την πρόσδεση των εμπορευματοκιβωτίων αλλά και με το υπέρβαρο αυτών συχνά. Ε, κάποιες φορές έχει να κάνει και με την ηλικία του σκάφους, με, το μέγεθος του σκάφους, όπως είπε ο κύριος ε, Higgins. Η ασφάλεια και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως είπα και, νωρί... και πριν, είναι πολύ σημαντικό και είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν. Δεν μπορούμε να συμβαστούμε σε αυτά τα θέματα και και εγώ και ο Αντιπρόεδρος Κάλλας θα εξετάσουμε την, ε, το ενδεχόμενο περαιτέρω δράσης και θα συνεργαστούμε εκ του σύνεγγυς μαζί σας και με την Επιτροπή σας κύριε Σίμψον ούτως ώστε να προχωρήσουμε. Ε, έχουμε ήδη αρκετά εργαλεία στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την πρόληψη της ε, ρήπανσης και από τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα. Τώρα, για τη συγκεκριμένη δράση που πρέπει να αναλάβουμε, σε αυτή τη φάση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να δράσουμε. Παρότι καταλαβαίνω ότι εσείς θεωρείτε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακό Οργανισμός είναι πολύ αργοκίνητο και ότι η Κομισιόν θα πρέπει να πιέσει για πιο γρήγορε λύσει. Ε, ξέρω ότι ο Αντιπρόεδρος Κάλλας ε, πιστεύει ότι η κατάλληλη μορφή, ο κατάλληλος χώρος για να συζητήθει αυτό το θέμα είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και μια αναθεώρηση του προγράμματος για, ε, την πρόθεση στη θάλασσα επιβεβαιώνει τη σημασία για μια παγκόσμια προσέγγιση, ούτω ώστε να έχουμε και διαδικασίε και, πρότυπα, ούτω ώστε ε, όλα τα πλοία και από τα κράτη-μέλη και από άλλα κράτη να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Κλείνοντα, θέλω να τονίσω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει καταρχήν να συζητηθεί στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που συμμετέχει η Κομισιόν ω παρατηρητή και ετοιμάζουμε μάλιστα ω Κομισιόν τη θέση μα ε, μαζί με τα κράτη-μέλη. Σας διαβεβαιώ ότι θα διαβιβάσω τα αποτελέσματα της συζήτηση ε, στον Αντιπρόεδρο Κάλλας και ξέρω ότι δεν θα μελήσει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μάσνερ. Ολοκληρώθηκε εδώ πέρα η συζήτηση. Περνάμε τώρα στην έκθεση της ε, Τώρα στην έκθεση κυρία Μάισνερ για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Τον λόγο λοιπόν έχει η συγγήτρια για